προηγουμένως. Τώρα α ηρεμήσουμε και α περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρα διάταξη που είναι η κοινή συζήτηση Συμφωνία Εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Σιγκαπούρη. Η συζήτηση θα γίνει από τη βάση της έκθεσης του David Μάρτιν για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης. Επιπλέον έχουμε ένα ψήφισμα και μια σύσταση που αφορά την προστασία των επενδύσεων μεταξύ των δύο. Και άλλη μια έκθεση του κύριου Μάρτιν και άλλο ένα ψήφισμα και μια σύσταση του κύριου Ιστούρης. και άλλη μια έκθεση του Αντώνιο Λόπεση Τούρι White Ω ψήφισμα για την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σιγκαπούρης. Ξεκινάμε τις συζητήσει. Καλώ ήρθατε κυρία Επίτροπε. Πρώτο ομιλητή. θα είναι ο εισηγητή, ο κύριο Ντέβιτ Μάρτιν. Ε, ναι. Very much. Επιτέλους, μετά από 10 χρόνια συζητήσεων βρισκόμαστε εδώ μετά από πολλά εμπόδια, πολλές τροφές. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση Σιγκαπούρης για την ε, υπομονή της και τον πρέσβη της Σιγκαπούρης για την καλή συνεργασία του. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την Γενική Διεύθυνση Trade για μια συμφωνία την οποία μπορούμε πιστεύω να στηρίξουμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και ηγητές για την πολύ καλή συνεργασία. Κάποιοι μπορεί να είναι ακόμα σκεπτικοί, στες, ε, τι δεν είναι καλό για ε, σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία βασίζεται στη συμφωνία με τον Καναδά και την Ιαπωνία. Στέλνει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη σε ένα σύστημα εμπορίου που θα βασίζεται σε κανόνε. Ενώ ο Ντόναλτ Τραμπ θέλει να στήσει τείχου και τείχη, εμεί του καταργούμε και δημιουργούμε ζώνες ελεύθερων συναλλαγών. Η Σιγκαπούρη είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για ε, το ευρωπαϊκό εμπόριο και τις επενδύσεις και τι, και τι καταφύγιο, ένα σημαντικό, μια σημαντική αγορά, μια χώρα που είναι προσιλωμένη στο κράτος δικαίου, ε, με ένα από τα υψηλότερα κατακεφαλή εισοδήματα στον κόσμο. Πάνω από 10.000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ε, την βάση τους εκεί. Και πολλές από αυτές, ε, με εργαλείο αυτή τη συμφωνία, θέλουν να διευρύνουν τι δραστηριότητε του στη Σιγκαπούρη μέσω, των, μέσω ε, εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι και στρατηγική σημασία χώρα η Σιγκαπούρη για να έχουμε πρόσβαση στην ε, ασιατική περιοχή, στην περιοχή αυτή της Ασίας, η οποία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ένα μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών μας προς την περιοχή αυτή περνούν ε, από τη Σιγκαπούρη. Και αν δεν κάνουμε τίποτα, δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη έχει ήδη εταιρική σχέση με τι χώρε του Ειρηνικού, θα μείνουμε πίσω. Από οικονομική πλευρά, είναι λοιπόν αμοιβαία ωφέλιμη αυτή η συμφωνία. Όμω επιπλέον των εμπορικών ωφελών, θα μπορούσα να πω ότι η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει σαφώ και τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ επίση και τι θέσει του Κοινοβουλίου που έχουν επαναληφθεί επανειλημμένω στο παρελθόν. Για παράδειγμα, τίποτα σε αυτή τη συμφωνία ε, δεν θα εμποδίσει την εφαρμογή της αρχή προφύλαξη προκειμένου κυβερνήσει να μοθετούν οι όφελο των πολιτών τους. Ε, προστατεύονται οι δημόσιες υπηρεσίες, ε, οι εισαγωγέ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ, προδιαγραφές, προσήλωση στην, προσήλωση, στην προστασία του περιβάλλοντος, της τη Γεωργία, και ε, προϋποθετήθεται η ε, σύναψη άλλων διεθνών συμφωνιών όπως η Συμφωνία του Παρισιού. Επίσης αναλαμβάνεται από τη Σιγκαπούρη η υποχρέωση να υπογράψει τις τρεις συμφωνίες του ΑΕΛΟ, της Διεθνούς Οργανωσής Εργασίας, που δεν έχει υπογράψει ακόμα. Ε, επίσης, ε, ε, αναλαμβάνουν την ευθύνη να δημιουργηθεί μια ομάδα, διαϋπουργική ομάδα προκειμένου να εφαρμοστούν αυτέ οι συμφωνίε σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Είναι η πιο προοδευτική επενδυτική συμφωνία που έχουμε διαπραγματευτεί μέχρι τώρα και θα πρέπει να αποτελέσει μοντέλο για το μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την όλη ομάδα της ε, για το ρόλο του στη διαπραγμάτευση προβλέπεται ένα μόνιμο ε, επενδυτικό δικαστήριο, έναν διοντολογικό κώδικα για τους δικαστές, ένα μηχανισμό έφεσης και ε, τη χρήση του πολυμερούς Διεθνούς Δικαστηρίου Ρυθμιστών Διαφορών. Αντικαθιστά τις 13 διμερείς σχέσεις προστασία των επενδύσεων που έχουν αυτή τη στιγμή κράτη-μέλη με τη Σιγκαπούρη. Υπάρχει μία δυναμία σε αυτή τη συμφωνία που θα πρέπει να καλυφθεί στις μελλοντικές συμφωνίες. Τους δίνει στου επενδυτέ δικαιώματα, αλλά όχι υποχρεώσεις. Με αυτή την επιφύλαξη μπορώ και τις δύο συμφωνίες να τις ε, συστήσω προς ψήφιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μάρτιν, λέει ο πρόεδρος. Έχω ένα αίτημα, έχουμε καθυστερήσει, είμαστε καθυστερημένοι για κατά 15 λεπτά. Παρακαλώ πολύ, ας παραμείνουμε ο καθένας στο χρόνο που του δίδεται για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση πριν τα μεσάνυχτα. Οπότε δεν θα κάνω δεχτέ τι μπλε κάρτε. Ο άλλος εισηγητή, ο κ. Λόπεθ, Ιστούρη Σουάιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Ντέβιτ Μάρτιν. Θέλω και εγώ να συγχαρώ, να ευχαριστήσω τον πρέσβη της Σιγκαπούρης. Μας βοήθησε πάρα πολύ ε, στην επεξεργασία αυτών των νομοδοτήσεων, των εκθέσεων. Ε, μας έδωσε με διαφανή τρόπο πολλές πληροφορίες για τη Σιγκαπούρη. 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε, που μάλλον το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Εδώ τελειώνει η διαδικασία αυτή. Αύριο θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα με την ψηφοφορία. Ε, προκειμένου να συμφωνήσουμε με το πλαίσιο συνεργασίας και τις συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων ε, των επενδυτών. Μία ακόμα φορά στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολυμερή διεθνή συνεργασία σε θέματα εμπορίου, αντίθετα με άλλους. Σε αυτή τη στιγμή αυτή η πολυμερή προσέγγιση τίθεται υπό αμφισβήτηση. Εμείς επιμένουμε στη διεθνή συνεργασία. Αυτή η συμφωνία προσπαθεί να θεσμοθετήσει Σχέσει σχέσεις οι οποίες υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες βασίζονται σε μακρά ιστορία φιλίας και οικονομικούς, ε, κοινωνικούς και πολιτικούς δεσμούς. Ε, θα αποτελέσει ένα νομικό πλαίσιο για την συνεργασία μεταξύ Σιγκαπούρ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Στόχος είναι η συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης, ασφάλειας, κλιματικής αλλαγής και ανάπτυξης μεταξύ άλλων. Ε, πράγματα τα οποία στα οποία δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι πολίτες μας. Η Σιγκαπούρη είναι σημαντικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η περιφερειακή ισορροπία στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Κάτι που είναι σημαντικό για την Ευρώπη, για τις επιχειρήσεις μας και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Σιγκαπούρη είναι η πόρτα εισόδου στην ασιατική αγορά και μια πλατφόρμα για τι ε, ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη κοντά στην Ιαπωνία, την Κίνα και άλλε οικονομίε, σημαντικέ οικονομίε τη περιοχή. Η συμφωνία αυτή θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στου Ευρωπαίου επενδυτέ. Να υπογραμμίσω ότι στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία θα δημιουργηθεί μια μόνη μεικτή επιτροπή με αντιπροσώπου των δύο πλευρών σε υψηλό επίπεδο έτσι ώστε καθημερινά να εργάζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι συνεργασία. Θα Είμαστε σημαντικοί συνομιλητέ σε θέματα που θα έχουν σχέση με την διεθνή ασφάλεια, την συνεργασία σε τεχνολογικό, ερευνητικό επίπεδο, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και τις μεταφορές, ιδιαίτερα τις θαλάσσιες και αέριες μεταφορές. Θα συνεργαστούμε σε θέματα ε, πληροφορίας ε, ε, και ανταλλαγής πληροφοριών. Οι επιχειρήσεις μας αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, χάνουν πολλά εκατομμύρια από κυβερνοεπιθέσεις, τις οποίες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνεργασία. Πολιστικές ανταλλαγές ήδη υπάρχουν, θα τις διευρύνουμε. Προγράμματα όπως το Μούντι και το Εράσμους ε, θα διευρυθούν και θα εφαρμοστούν και για τη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη μπορεί να γίνει πλατφόρμα ε, για τους νέους μας προς τις χώρες της ε, Ασίας. Επίσης, είναι σημαντική για τη συνολική παγκόσμια ασφάλιση και την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Χρειαζόμαστε γέφυρες συνεργασίες με τις άλλες χώρες, ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ε, μείωση της χρηματοδότησης ε, και γενικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία αυτή θα είναι πολύ καλή λοιπόν και για τους επιχειρηματές και για τις επιχειρήσεις ε, για να δημιουργήσουν σχέσεις όχι μόνο με τη Σιγκαπούρη αλλά και με άλλους χώρες της Ασίας. Πάνω από 10.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες βρίσκονται ήδη στη Σιγκαπούρη, την χρησιμοποιούν ως κέντρο για να εξυπηρετήσουν όλη την περιοχή του Ειρηνικού. Ένα μόνιμο νομικό πλαίσιο θα αποτελέσει ακρογωνίο λίθο της συνεργασίας μας και θα δώσει νομική ασφάλεια σε επιχειρήσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε καινούριε ευκαιρίε εμπορίου, προάγουμε τι επενδύσει, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή του. Κάθε φορά που οι πολίτε μα μπορούν να αναπτύσσουν τι ιδέε του και τα σχέδιά τους με τρόπο ασφαλή σημαίνει ότι δημιουργούμε καινούριες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Το είπα και πριν και θέλω να το επαναλάβω. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η σημαντική γεωπολιτική θέση της Σιγκαπούρης για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση κλιματικών ε, φαινομένων στην όλη περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας η Σιγκαπούρη θα μπορέσει να βοηθήσει ε, και ε, μάλλον εμεί θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Σιγκαπούρη στην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων που έχει πάρει για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, γιατί έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Τέλο, να ευχαριστήσω του και ηγητέ για τη βοήθειά του, για τη συνεργασία του και ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε με ευρία πλειοψηφία να ε, ψηφίσουμε και να εγκρίνουμε αυτό το πλαίσιο συνεργασία με τη Σιγκαπούρη. Είναι επιτυχία και επίτευγμα για όλους μας, ε, καθώς επίσης και ε, σημαντική πηγή σταθερότητας ε, και θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να μιλάτε μία φωνή. Τώρα η κυρία Μάλμστρομ, εξ των Κομισιόν. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Να ευχαριστήσω του δύο εισηγητέ, τον κύριο Ντέβιν Μάρτιν και τον κύριο Λόπε Ιστούρι Βουάιτ για τη δουλειά που έχετε κάνει και την καινή σα πόρια που μα έφερε σήμερα εδώ. Λίγα μέρη συμβολίζουν τα πλεονεκτήματα του εμπορίου και των επενδύσεων όσο η Σιγκαπούρη, η οποία έχει ε, επιδείξει ένα ανοιχτό πνεύμα, μια παγκοσμιοποίηση και έχει μεταμορφωθεί χωρίς φυσικούς πόρους σε μια της πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη έχει γίνει υπόδειγμα οικονομικού μετασχηματισμού και χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το εμπόριο, επενδύσεις, οι, βιώσιμες, ε, η βιώσιμη ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι. Και βεβαίως η ίδια αντίληψη ε, έχει ωφελήσει και εμάς στο παρελθόν και πρέπει να μας καθοδηγεί και στο μέλλον. Στενή εταίρη, εδώ και δεκαετίε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σιγκαπούρη αποφάσισαν να επισφραγίσουν την ε, συνεργασία τους μέσω των τριών αυτών συμφωνιών. Η νέα αυτή συμφωνία θα θέσει το γενικότερο πλαίσιο της ε, διμερούς συνεργασίας, πολιτικής συνεργασίας αλλά επίσης είμαστε και πολύ στενοί εταίροι εμπορίου και επενδύσεων. Είναι ο μεγαλύτερος μας εταίρος στην Ανατολική Ασία και στους 20 ε, κορυφαίους επενδυτές για αγαθά, στους 5 κορυφαίους ε, στις ε, επενδύσεις και από τους 10 κορυφαίους στο εμπόριο. Και έτσι θα αναπτυχθούν περισσότερο αυτοί οι δεσμοί τα ωφέλη είναι πολλά. Οι δασμοί στο διμερές εμπόριο θα καταργηθούν. Τα μη δασμολογικά φράγματα για ευρωπαϊκές εξαγωγές ε, επίσης ε, θα καταργηθούν. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, δημόσιες προμήθειας θα βελτιωθεί. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και για τους ανθρώπους και τις δύο πλευρές. Επίσης υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά το εμπόριο και την ανάπτυξη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, το περιβάλλον, την βιοπικιλότητα, την οικολογική σήμανση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και πότε ένα σημαντικό ρόλο στις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών της Σιγκαπούρης. Η κύρωση και η συμμόρφωση με τις ε, συμβάσεις του ILO θα είναι από τα πρώτα σημεία τα οποία θα παρακολουθήσουμε και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ε, μέχρι να τεθεί ενισχύση. Και ήδη οι αρχές Σιγκαπούρης ε, προετοιμάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την αηφόρο ανάπτυξη. Επίσης αυτά τα έχουμε διαπραγματευτεί σε συνδυασμό με μια συμφωνία για προστασία των επενδύσεων που έχει αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την οποία συνδιαμόρφωσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ. Το σύστημα αυτό αντιμετωπίζει τις ανησυχίες κοινωνία των πολιτών για ασαφείς κανόνες, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη δυνατότητας ε, προσφυγής, ε, έλλειψη ανεξαρτησίας ε, των επιδιαιτητών. Οπότε, με βάση την διαπραγματευτική μας εντολή, σας παρουσιάζουμε μια συμφωνία η οποία καθιστά πιο αυστηρές αυτές τις προδιαγραφές για να μην υπάρξει κατάχρηση. Μια συμφωνία η οποία πλήρως σέβεται τα δικαιώματα των κυβερνήσεων να φέρουν νέα νομοθεσία για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και άλλων δημοσίων αγαθών και δημιουργεί ένα πλήρως διάφανο σύστημα δικαστηρίων, κάτι το οποίο και ο Γενικός Αγγελέας ε, θεώρησε πλήρως συμβατό με τις συνθήκες ε, στην περίπτωση της συμφωνίας με τον Καναδά και θα μπορούσαμε έτσι να καλύψουμε και τις υφιστάμενες 3.000 εμπορικές συμφωνίες ε, παγκοσμίω. Και θα έχουμε έτσι μια εξέλιξη για να έχουμε και υποχρεώσεις των επενδυτών όπως ανέφερε ο κύριος Μάρτιν. Οπότε οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες που είναι πραγματικά η τελευταία λέξη των συμφωνιών αυτών και βεβαίως η Σιγκαπούρη είναι η καρδιά του εμπορίου της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει η συμφωνία αυτή ε, υπόδειγμα και για τους άλλους εταίρους. Και τέλος, ε, για την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για εμά και τη Σιγκαπούρη, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Παρέχει μια βάση, όπω είπε ο εισηγητή, για αποτελεσματικέ διμερείς σχέσει με τη Σιγκαπούρη, για ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και για ενίσχυση τη συνεργασία σε πολλούς τομείς. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, δικαιοσύνη, ασφάλεια, συνδεσιμότητα, διαπροσωπικές επαφές, ε, πληροφορική, πολιτιστικές ανταλλαγές, αλλά και απασχόληση και κοινωνικά. και θα μας επιτρέψει να εντείνουμε τις συνεργασίες σε τομείς όπως η ενέργεια, του περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η προστασία των ψυχών πόρων, έξυπνες πόλεις και μεταφορές. Και βεβαίως σε περίπτωση διαφωνιών θα συσταθεί μια διμερής επιτροπή υψηλού επίπεδου για την ορθή λειτουργία και εφαρμογή της ε, συμφωνίας αυτής και βεβαίως ε, θα προστατεύσουμε και τους στόχους της για την ε, περιφερειακή δυναμική. Η Σιγκαπούρη μας έχει επιδείξει πως ε, είναι υπέρ ε, της πολυμερούς προσέγγισης στην Νοτιοανατολική Ασία και εκτιμούμε ιδιαίτερο την συνεργασία μας και θα φροντίσουμε να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Η συνεργασία με την Σιγκαπούρη για ζητήματα που αφορούν τον Αζίαν είναι πολύ επικοδομητική μέχρι στιγμή. Οπότε η συνεργασία των δύο μερών είναι βαθιά και ευρύτατη ήδη σήμερα και δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οι δυνατότητε για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία είναι μεγάλες. Με βάση ένα κοινό όραμα, ένα πολυμερές σύστημα που θα βασίζεται σε κανόνες. Να ευχαριστήσω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένουμε την στήριξή σας στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η αρχή της συζήτησης είναι πολλά υποσχόμενη, πολύ διαφορετικός ο τόνος από ό,τι στην προηγούμενη. Ο κύριος Κέλλη για το ΕΛΚ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές. Πολύ καλή συνεργασία σε αυτό το θέμα και τους δύο εισηγητές θέλω να ευχαριστήσω. Καθυστέρησαν πολύ, αλλά ευτυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος. Ελπίζω αύριο να ψηφίσουμε και να το εγκρίνουμε. Το εμπόριο ανάμεσα στην Καπορ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 55 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 44 δισεκατομμύρια εξαγωγέ τη Σιγκαπούρη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνονται πολύ γρήγορα αυτά τα νούμερα έτσι κι αλλιώ. Είναι πολύ καλή λοιπόν αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Συγχαίρω την κυρία Μάλστρομ για την πολύ καλή δουλειά τη. Ε, θα ωφεληθούν πολλοί κλάδοι. Ο πολιτικό κλάδο, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, όπω ξέρω. Αυτή η συμφωνία δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί για όλους, προς όφελος όλων. Με την απόσυρση των εμπορικών φραγμών, δασμολογικών και μη δασμολογικών, ε, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Το πολυμερές δημοσιονομικό ε, δικαστήριο είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και ε, μετά την αν συμφωνήσαμε στις συμφωνίες με τον Καναδά και την Ιαπωνία, σίγουρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε και εδώ και μακάρι αύριο με λίγο Ιρλανδέζικο whisky να το γιορτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Θα μπορούσατε να σέβεστε λίγο το χρονικό όριο, το χρόνο που σας δίνουμε. Κυρία Μαρία Μόσκα. Επίτροπε, συνάδελφοι, λίγε εβδομάδε πριν την ψηφοφορία, ε, λίγε εβδομάδε μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου αυτού για τη συμφωνία με την Ιαπωνία, πάλι μιλάμε για τη σύναψη στρατηγική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πολίτε τη, του εργαζομένου τη και τι επιχειρήσει τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ψηφοφορία ε, που δεν έγινε για τη συμφωνία με τι ΗΠΑ τώρα θέλει να γίνει πρωταγωνιστής στο διεθνέ εμπορικό προσκήνιο. Η τρίτη οδός για το εμπόριο που θέλει να αντιμετωπίσει τον άκρατο ανταγωνισμό και τον ανεξέλεγκτο φιλελευθερισμό ποτέ δεν ήταν τόσο ελκυστική. Θα πρέπει να προβάλλουμε τι προδιαγραφέ και τα πρότυπά μα σε διεθνές επίπεδο. Χάρη στι ρήτρε για την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώ και του περιβάλλοντο, θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε και του πολίτε από τι παράπλευρε συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση. Για να αναφέρω μερικά, η δεσμεύσει τη Σιγκαπούρη για την κύρωση των συμβάσεων του ILO, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία, για τον σεβασμό τη Συμφωνία ε, για το Κλίμα των Παρισίων, καθώ και την αναγνώριση των γεωγραφικών μα ενδείξεων, όπω η προστατευόμενη προέλευση και η προστατευόμενη καταγωγή. Εδώ θα, γεωγραφική ένδειξη, μάλλον. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια με την τέταρτη οικονομική δύναμη σε ανάπτυξη ε, και πώ θα φτάσουν τα προϊόντα στα σύνορά μα. Είναι μια σημαντική διέξοδο για να στηρίξουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη ανάπτυξη. Η Σιγκαπούρη είναι μια ανοιχτή πόρτα για την ε, Νοτιοανατολική Ασία, τι χώρε Αζεάν. Είναι η πιο δυναμική οικονομία του κόσμου. Είναι η έβδομη σε σημασία χώρα για τι εξαγωγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 30% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που έχουν παρουσιαστεί στην Σιγκαπούρη είναι μικρομεσαίες και οι εξαγωγές έφεραν κέρδη 33 δις ευρώ στις επιχειρήσει μα. Η συμφωνία θα επιτρέψει να πολλαπλασιαστούν τα νούμερα αυτά και θα δημιουργήσει πολλαπλέ θέσει εργασία στην Ευρώπη χωρί κανένα κόστο. Η βιομηχανία στη Σιγκαπούρη είναι συμπληρωματική προ την Ευρωπαϊκή. Στον βιομηχανικό κλάδο αλλά και στη Γεωργία δεν υπάρχει κανένα κομμάτι τη οικονομία μα που δεν θα ωφεληθεί από τη συνεργασία με τη Σιγκαπούρη. Σε σχέση με τα γεγονότα αυτά και τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίε. Οι συμφωνίε αυτέ είναι καθοριστική σημασία για του εργαζομένου τη Ευρώπη. Τα προϊόντα μα και τα αγαθά μα πολλούνται και ε, εκτιμώνται σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στη συμφωνία αυτή, περιορίζοντα τι αρνητικέ πράγματα συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρου του ECR, ο κ. Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, η Συμφωνία Ελεύθερη Συνεργασία με τη Σιγκαπούρη είναι ένα ακόμα παράδειγμα τη ε, ε, επιτυχημένη εφαρμογή ε, το, ανοίγματο των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την Ιαπωνία, για παράδειγμα, ανοίγουν αγορέ και άλλε αγορέ. Ε, η Βρετανία βρίσκεται 45 μέρε πριν την ε, αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αλλά να σας θυμίσω όλα αυτά τα οποία, τα ψευδή τα οποία είχαν υποσχεθεί οι υπέρμαχοι του Brexit την, ε, για, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι υποσχόντουσαν, υποσχόντουσαν ότι η, η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ενδιαφερόταν ούτε μπορούσε να συνάψει συμφωνίες που να ωφελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να όμως που βλέπουμε μια τέτοια συμφωνία ε, που έρχεται κατόπιν το συμφωνία του Καναδά, την Αυστραλία και, την και και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ οι συμφωνίε με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είναι επίση πολύ προχωρημένε. Είναι προφανέ πλέον ότι μετά τι 29 Μαρτίου οι 27 χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πολύ περισσότερε ευκαιρίε να κάνουν εμπόριο με τη Σιγκαπούρη από το Ηνωμένο Βασίλειο για τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Τάισον, ε, επιχειρηματία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέρ του Brexit, ε, έχει ήδη ξεκινήσει να χτίζει ένα εργοστάσιο για ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Σιγκαπούρη και μετέφερε την έδρα του από τη Βρετανία εκεί. Τι άλλο να πω, ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ΑΛΔΕ, ο κ. Θερμός Εμπαλσέλς. Αγαπητέ κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η συνεργασία ανάμεσα στον David Μάρτκιν και τους και ηγητές ήταν εξαιρετική και γι' αυτό το λόγο είχαμε ε, μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Επίσης να ευχαριστήσω τον πρέσβη Σιγκαπούρης και την κυβέρνηση Σιγκαπούρης για την ε, υπομονή τους στηρίζω και την Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών και το Μηχανισμό προστασία Επενδύσεων. Είναι αμοιβαία ωφελός ε, αμοιβαίω ωφελή ε, συνεργασία και για τη Σιγκαπούρη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εταιρείε του. Οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν το 2009, Δεκέμβρη 2009. Σχεδόν 10 χρόνια μετά βρισκόμαστε στο τέλο του δρόμου αυτού. Ε, είναι ο, ο μεγαλύτερος ε, εταίρος μας στην περιοχή, ε, πάνω από 10.000 ε, ευρωπαϊκέ εταιρείε έχουν τα περιφερειακά του γραφεία στην Καπούρη και ε, δρούν σε ένα αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον. Είναι επίσης ε, κόμβο για όλη την Ασία Σιγκαπούρη, μεταφορικός και εμπορικό. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο και για τι άλλε ασιατικέ χώρε. Είναι η πρώτη σε αυτή την περιοχή που υπογράφουμε. η συμφωνία Προστασία των επενδύσεων αντικαθιστά 13 διμερείς αντίστοιχε συμφωνίε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ κρατών μελών και τη Σιγκαπούρη. Αύριο ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε αυτό, αυτό το νέο, μοντέρνο σύστημα προστασία επενδύσεων που θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε τους θεμητούς στόχους της εμπορικής μας πολιτικής δίνοντας ε, ασφάλεια και προστατεύοντας το περιβάλλον. Επίσης, ε, η συμφωνία αυτή ορίζει μια μεταχείριση των εταιριών χωρίς διακρίσεις ε, και ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Θα ήθελα τέλος να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω την κυρία Μάλστρομ για τις προσπάθειές της. Ε, μας βοήθησε πάρα πολύ σε πλήρη διαφάνεια. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη έρχεται με το εμπόριο, κυρίε και κύριοι, όχι με μεγαλύτερα κρατικά χρέη. Με τον Brexit και τον Τραμπ ο, η πολυμερής προσέγγιση κινδυνεύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα, εξ ονόματος ε, της ε, Γκουε, η κυρία Αν Μαρή Κύριε Πρόεδρε, έχω τρεις σοβαρές επιφυλάξεις για αυτήν τη συμφωνία. Περιλαμβάνεται πάλι μια παραγραφός για το ISDS, δηλαδή κάποιο διαιτητικό δικαστήριο για τους επενδυτές. Αυτό είναι κατ' ουσίαν. Γνωρίζουμε πως εδώ πέρα έχουν δικούς τους κανόνες οι επιχειρήσεις και μπορούν να σέρνουν τα κράτη ενώπιον αυτού του δικαστηρίου και να πληρώνει ο φορολογούμενος. Εδώ πέρα υπονομεύεται το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Δεύτερον, η σύμβαση προσφέρει αποκλειστικά δικαιώματα σε επενδυτές, αλλά δεν υπάρχουν κανόνες υποχρεωτικοί για την υλοποίηση των διατάξεων περιφορίας. Εδώ πέρα λοιπόν θα υποφέρουν άνθρωποι, ζώα και περιβάλλον. Τρίτον, υπάρχει ρητά η δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να αγοράσουν κρατικά ομόλογα και σε καιρούς κρίσης μπορούν να προχωρήσουν σε να μπλοκάρουν, συγχωρείτε, αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους το Κοινοβούλιο και οι Κομισιόν εδώ πέρα υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα πολυεθνικών επενδυτών και τα βάζουν πάνω από το συμφέρον των πολιτών. Είναι απαράδεκτο. Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψαν μια αίτηση κατά του ISDS ακριβώς για να σταματήσουν τέτοιες συμβάσεις. Σταματήστε λοιπόν το ISDS, σταματήστε αυτήν την εμπορική συνθήκη και σταματήστε την ταξική δικαιοσύνη για τις πολυεθνικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για τους πράσινους ο κύριος Μπιουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, λέμε, στην ε, Γερμανία. Και βεβαίως άργησε πολύ. Και πρέπει να πω ότι ήταν πολύ υπομονετική η Σιγκαπούρη και την συγχαίρω ακριβώς για το ότι βοήθησαν στον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αζίαν. Η συμφωνία δείχνει ότι η Ευρώπη επιθυμεί την ενισχυμένη συνεργασία με τον Αζίαν για το συμφέρον μας και για τις αξίες μας. Χρειαζόμαστε στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις και χρειαζόμαστε μια τέτοια σχέση με τον Αζίαν για να προωθήσουμε την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού και θέλουμε και πολυμερή συνεργασία και τέλος θέλουμε την πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ελευθερία του συνέρχεστε μέχρι την κατάληξη θανατικής ποινής. Αλλά επίσης πρέπει να θέσω ένα πρόβλημα και το λέω στα αγγλικά για να γίνει αντιληπτό και στην Σιγκαπούρη. Τα ομόλογα, δεν, τα κρατικά ομόλογα δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τις συμφωνίες προστασίας των επενδυτών. Από την κρίση του 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες ε, διαδικασίες για την αναδιάρθρωση χρέους σε περίπτωση χρεοκοπίας. Εδώ πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα παραθυράκι με τη Συμφωνία της Σιγκαπούρης. Όπως λέει και η Handelsblatt ε, σήμερα, η συμφωνία αυτή αυξάνει το κατόφλι για την συνένεση των πενητών σε περίπτωση αναδιάρθρωσης χρέους σε σχέση με το επίπεδο που ισχύει αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επενδυτέ ε, που λειτουργούν με βάση αυτήν τη συμφωνία έχουν προνόμια σχέση με άλλου επενδυτέ και αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό απαιτούμε η συμφωνία αυτή να μην ψηφιστεί αύριο μέχρι να καταργηθεί το περάρτημα 4 και το δημόσιο χρέος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μιλάτε χωρίς να σας δώσω το λόγο. Συνάδελφε, στο έδρανο 39. Σας παρακαλώ. Ωραία. Εκ μέρους του FTD. κυρία Μπεκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε στις πολυεθνικές να κάνουν τη δουλειά των κρατών. Σε αυτό το κοινοβούλιο φαίνεται ε, ότι όλοι συμμετέχουμε τον ίδιο τρόπο, αλλά και εσείς ε, εκπροσωπείτε με τον ίδιο τρόπο τους πολίτες, υποτίθεται. Δεν μπορείτε λοιπόν να βάλετε αποφάσεις σε αυτή τη σύνοδο χωρίς να είναι πραγματικά ανεξάρτητες. Δεν μπορεί να ψηφίζετε υπέρ μια συμφωνία για επενδύσεις με τη Σιγκαπούρη. Και είναι ακόμη χειρότερη η συμφωνία αυτή από τη ΣΕΤΑ. Οι πολυεθνικέ ουσιαστικά θα έχουν υποχείριο τις χώρες μας ε, τι κυβερνήσει, τι περιφέρειες, του αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση. θα μπορούν από δικαστήρια επίλυση διαφορών επενδυτών κρατών να διαλυθούν τα κράτη, να ε, είναι θύματα των επενδυτών. Εγώ πιστεύω στο παγκόσμιο εμπόριο και πάντοτε το υποστηρίζω όταν μιλάμε για συγκεκριμένα κέρδη και ωφέλη για τι επιχειρήσει μα. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για εμπόριο, μιλάμε για συμφωνίε άλλου είδου και πρέπει να γίνει μια σαφή διάκριση. Υπάρχει συμφωνία για τι επενδύσει, που θα επιτρέψει τι πολυεθνικέ να ε, αποδηγετήσουν ουσιαστικά τα κράτη, αλλά υπάρχει και το θέμα των συναλλαγών, που αφορά μόνο τι εξαγωγέ και τι εισαγωγέ. Αυτή η διάσταση εισαγωγών-εξαγωγών είναι σίγουρα θετική για την ε, οικονομία μα. Θα μα επιτρέψει να αναπτυχθούμε σε μια νέα αγορά που θα εκμεταλλευτεί και την ανάπτυξη τη Αυστρία. Ε, τη Ασία, συγγνώμη. Εδώ όμω δεν χρειαζόμαστε μια τέτοια συμφωνία. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι διαπραγματεύσει αυτέ ε, εκπονήθηκαν με έλλειψη διαφάνεια και να πω ότι η Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο μόνα για πράγματα που ήδη ήταν τετελεσμένα γεγονότα και για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων κυρίω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα κοιτάξουμε με ιδιαίτερη προφυλακτικότητα το πώ θα αντιδράσουμε στην ψήφιση αυτή τη συμφωνία. Και υπάρχει και το θέμα των επενδύσεων. Η συμφωνία για, ε, για τι επενδύσει περιέχει αυτή τη ρήτρα για την περιβόητη επίλυση των διαφορών και το σχετικό όργανο δικαστήριο. Είχαμε αντιταχθεί ε, έντονα και σφοδρά και στην ανάλογη διάταξη στη Συμφωνία ΣΕΤΑ και γι' αυτό μα έχουν ψηφίσει πολίτε για να καταψηφίζουμε τέτοιου είδου ιδέε. Ευχαριστούμε και τώρα ε, για την ΕΝΕΦ e ο κύριο Ζαμέ. Η κυρία Ζαμέ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, εδώ το εμπόριο σίγουρα δεν ε, έχει δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια, αλλά αυτό είναι το κρέντο, το πιστεύω των ε, γραφειοκρατών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταργώντα τα σύνορα, η συμφωνία με τη Σιγκαπούρη θα μα κάνει αποθήκη και ε, σταυροδρόμι του παγκόσμιου εμπορίου και θα προσθεθεί η συμφωνία αυτή σε όλες τις υπόλοιπε. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτε μα στα εμπορεύματα τη Ασία, του Ειρηνικού, τη Νότια Αμερική. Κάτι που σίγουρα θα θέσει εναφιφόρο τη δική μα την οικονομία. Η συμφωνία αυτή μάλιστα είναι άκρο επικίνδυνη για του Γάλλου καταναλωτέ και του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Γιατί η Σιγκαπούρη δεν αναγνωρίζει ένα μεγάλο μέρο των γεωγραφικών μα ενδείξεων ε, και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ αξίε, να μην τι αναφέρω καν. Θα ήταν ε, κάτι που εκεί συστηματικά και ε, επανειλημμένω θα άρχιζαν τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Η, ελευθερία, η ελευθεροτυπία, τα δικαιώματα των ανθρώπων, οι γκρίζε ζώνε των φορολογικών παραδείσων. Τίποτα από αυτά δεν ενοχλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εμπόριο. Πάνω απ' όλα το εμπόριο. Αυτή η παγκόσμια επιδημία. Μόνο που ούτε η Γαλλία, ούτε η Ευρώπη δεν επωφελούνται από αυτέ τι συναλλαγέ των πολυεθνικών. Οι πολυεθνικές υποφελούνται σίγουρα. Πάντως αυτές οι, άκρατο, οι άκρατες φιλελεύθερες ε, πολιτικές είναι ουσιαστικά κοροϊδία τις οποίες δεν θέλουν άλλο οι λαοί. Θέλουν η παραγωγή να επιστρέψει στην επικράτειά τους. Τα προϊόντα να πηγαίνουν στις αγορές που μπορούν τα αγοράζουν εκείνη απευθεία και να τα βάζουν στο πιάτο τους. Αντιτασσόμεστα σε αυτή τη συμφωνία με αυτή την πολιτική παγκοσμιοποίηση των αγαθών Ευρωπαίων των μακάριων Ευρωπαίων. Αυτό που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να το αποδεχτεί και να το καταπιεί ο λαό. Σας ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην ε, κυρία Κβίστφουντ Ρόβολ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε κάποια σημεία μόνο. Πρώτον, ε, είναι η πρώτη συμφωνία που έρχεται μετά την απόφαση του ΔΕΚ για την αποκλειστική ή μεικτή αρμοδιότητα για τέτοιες συμφωνίες. Οπότε είναι μια σύγχρονη ε, συμφωνία αυτή την οποία θα ψηφίσουμε. Δύο σημεία τώρα. Το πρώτο κομμάτι της ε, συμφωνίας αυτής για τις ε, συμβάσεις του ILO. Η Σιγκαπούρη έχει δεσμευτεί γραπτός ότι θα τις κυρώσει. Ε, μα αυτό είναι αυτό που θέλουμε. Νομίζω ότι τελικά ε, είναι κάτι το οποίο είναι μια νίκη για εμάς και για την κυρία Επίτροπο για την προστασία των επενδύσεων. Έχουμε ένα διμερές δικαστήριο στο οποίο συμφωνήσαμε. Αυτό το οποίο δηλαδή ζητάμε εδώ και χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αναγνωριστεί γραπτός. Και αυτό θετικό για εμάς. Η Σιγκαπούρη θα μας ανοίξει την πόρτα για τις άλλες χώρες ε, του Αζίαν. Και αυτό θα το υπερψηφίσει ε, το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην κυρία Γκρας Βαντερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, η Κομισιόν μας λέει συνεχώς ότι θα έχουμε εμπόριο για όλους, αλλά πάλι δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Έχουμε μια ριζοσπαστική πολιτική της αγοράς, από την οποία κερδίζουν μόνο μεγάλες εταιρείε. Αηφορία, δικαιώματα εργαζομένων και περιβαλλοντικές προδιαγραφές περνάνε σε δεύτερη μοίρα, να μην πω ότι αγνοούνται εντελώ. Η Σιγκαπούρη δεν έχει κυρώσει τις 8 βασικές συμβάσεις του ILO. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κυρώσεων. Όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο κείμενο. Και το ICS βεβαίως είναι κάποια βελτίωση, αλλά το βασικό πρόβλημα δεν έχει παραμεριστεί. Οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν προνομιούχο θέση ε, και ξεπερνούν τα εθνικά δικαστήρια. Δεν είναι αυτό εμπόριο με βάση τους ε, κανόνες. Γι' αυτό θα καταψηφίσω και την εμπορική συμφωνία και την συμφωνία προστασίας ε, των επενδύσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάνν Ζάχραντιλ. Ευχαριστώ. Είναι η τρίτη μου θητεία σε αυτό το κοινοβούλιο. Και θυμάμαι πόσο κόπο χρειαστήκαμε και πόσο χρόνο χρειαστήκαμε να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ήδη είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία και μόλις τώρα ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας. Η Σιγκαπούρη είναι κόμβος για την Νοτιοανατολική Ασία και συνολικά για την Ασία. Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου διευρύνεται μετά τη συμφωνία με την Ιαπωνία στη συγκεκριμένη περιοχή. Και ετοιμάζουμε και άλλη μια παρόμοια συμφωνία με το Βιετνάμ. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε πριν τελειώσει η θητεία μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτρόπε, κυρίες και κύριοι. Τα αγαθά ανταλλάσσονται εδώ και αιώνες και σε μεγάλες αποστάσεις όσο είχαμε τρόπο να τα μεταφέρουμε. Τώρα όλο και περισσότερο εξαιτία τη ψηφιοποίηση και, και υπηρεσίε μπορούν να προσφερθούν. Ένας μεταφραστής από την Ασία μπορεί να μεταφράσει ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί εδώ. Για παράδειγμα. Οπότε εμείς δεν δημιουργούμε εμπόριο. Αυτό που κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίζουμε ότι οι κανόνες που το διέπουν ε, είναι προβλέψιμοι και δίκαιοι. Θέλουμε υψηλότερες προδιαγραφές και ε, να ωφελούμαστε όλοι. Ο, η και Τραμπ ε, δείχνουν τι μπορεί να προκληθεί από την έλλειψη κανόνων. Και είναι λίγο ηρωνικό το ότι επικρίνεται αυστηρά όχι τόσο το εμπόριο με την Κίνα για παράδειγμα, αλλά οι κανόνες εμπορίου που θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε μέσω των συμφωνιών. Οπότε χαίρομαι αυτούς που δείχνουν ότι είναι ηγέτες και τους εταίρους μας Σιγκαπούρη, με τους οποίους διαπραγματευόμαστε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Η Σιγκαπούρη είναι ένας μοντέρνος μίζων κόμβος στην περιοχή και ισχυρός μας εταίρος στην Νοτιοανατολική Ασία. Αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα καταστήσει Σιγκαπούρενους Ευρωπαίους, ούτε και εμείς θα τους αντιγράψουμε. Όπως πάντα είμαστε υπεύθυνοι εμείς για την νομοθέτηση των δικών μας κοινωνιών. Και χαίρομαι που βλέπω ότι πείσαμε τη Σιγκαπούρη να αντικαταστήσει τις 13 πεπαλαιωμένες πλέον διμερείς συμφωνίες επενδύσεων ε, που έχει με κράτη-μέλη ε, και να ε, συμφωνήσει με την δημιουργία του καινούριου μηχανισμού προστασίας επενδύσεων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πρώτο βάθμιο δικαστήριο και δεύτερο βάθμιο δικαστήριο. Αυτοί που δεν συμφωνούν με την ISDS, με το μηχανισμό επίλυση διαφορών, ε, θα πρέπει να είναι χαρούμενοι με αυτό το μοντέλο. Σε μια εποχή που ο προστατευτισμός, ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός ε, δείχνουν άνοδο, είναι σημαντικό να δώσουμε το χέρι στους εταίρους μας ε, στο πλαίσιο τέτοιων συμφωνιών που βασίζονται σε κανόνες δίκαιους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μορέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών ε, ε, διαδέχονται μια την άλλη και μοιάζουν. Ε, σε επιτάχυνση, σχεδόν ε, σε φρενήρια, μια και είμαστε το τέλο τη θετία, και μοιάζουν γιατί εξυπηρετούν κυρίω τα συμφέροντα όσων κατέχουν το κεφάλαιο ή των ε, ιδιοκτητών των πολυεθνικών, ει βάρο των μισθωτών και των εργαζομένων. Τίποτα το καινούργιο και σε αυτή τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Δεν υπάρχουν περιορισμοί και απαιτήσει στα περιβαλλοντικά πρότυπα, σε όσε ρήτρε ουσιαστικά θα ευνοούν τι τις επιχειρήσεις ε, εις βάρος των κρατών, ούτε κάτι για τις επενδύσεις. Εδώ όμως ε, θέλω να πω ότι οι ομόλογοι της Συγκαπούρης μας είπαν ότι έχουμε πολλές κοινέ αξίες με τις Ευρώπες. Μα δεν είναι καμιά ειρηνική κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι ένα πολυτεχνικό καθεστώς η Συγκαπούρη. Επίσης, για μας πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε την, ε, την αντίφαση αυτή. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής των φορολογικών παραδείσων, της αδιαφάνειας τα χρηματοοικονομικά. Από τη μια λοιπόν λέμε ότι θα ε, κυνηγάμε την ε, φοροδιαφυγή τη πάτε και από την άλλη με χαρά και σε τέτοια ψυχική εφορία θα εγκρίνουμε τέτοιε είδου συμφωνίε. Λέτε ότι είναι καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσαμε να έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο και πολύ κουπί. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριο Ζαντό, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, ε, είπατε ότι είναι πολλά τα, οφ, ε, τα οικονομικά οι οικονομικέ δυνατότητε τη Σιγκαπούρη και ότι είναι υπόδειγμα. Όμω δεν μιλήσατε καθόλου για την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία. Αυτό δεν το αναφέρατε καν. Και δικαίω. Γιατί αυτή η συμφωνία επενδύσεων ουσιαστικά τι κάνει, ε, δεν ε, λαμβάνει καν υπόψη ότι δεν υπάρχει δημοκρατικό καθεστώ. Δεν βλέπετε ότι αναπτύσσονται οι εθνικισμοί, οι λαϊκισμοί. Δεν βλέπετε ότι όλα αυτά υποδαβλίζονται, ότι καλλιεργούνται από την ε, άρνηση τη εθνική κυριαρχία που οργανώνει οργανώνεται διαρκώ και την ενισχύεται ει βάρο των πολιτών. Το βλέπουν αυτό και ωφελείται τι πολυεθνικέ. Είναι δεκάδε οι πολυεθνικέ που έχουν έδρα στην ε, Σιγκαπούρη και θα επιτεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία, το περιβάλλον, τι δημόσιε υπηρεσίε. Τώρα και για την αναδιάρθρωση του χρέου. Αυτό υπονομεύει τη δημοκρατία. Η Ευρώπη σημαίνει δημοκρατία. Η Ευρώπη θέλει του πολίτε τη. Δεν μπορεί να είναι για τι πολυεθνικέ. Επιτέλου, παρακαλώ, συνάδελφοι, απορρίψτε τη συμφωνία αυτή. Συλλήβδην. Δεν μπορούμε διαρκώ να υποστηρίζουμε τι πολυεθνικέ. Δεν μπορούμε διαρκώ να υποστηρίζουμε του φορολογικού παραδείσου και τα πολυτερχιά καθεστώτα. Αυτό υπονομεύει την δημοκρατία και καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σα ήταν σαφέ. Και τώρα... Ο Earl of Dartmouth. Ναι, Πολύ καλό που κάποιοι και κάποιο άλλο ε, δείχνει τέτοιο πάθο. Η Σιγκαπούρη είναι μια επιτυχημένη ιστορία. Μια ιστορία επιτυχία. Έχει υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ από την ίδια τη Γερμανία. Αλλά η Σιγκαπούρη, επαναλαμβάνω, ε, δεν είναι, δεν είναι, επαναλαμβάνω, ένα τμήμα, τμήμα ενός μεγάλου εμπορικού ε, σχηματισμού. Και αυτοί που θέλουν η Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το έχουν υπόψη τους. Και να απαντήσω στο προηγούμενο σχόλιο που έγινε. 45 χρόνια μετά την ένταξη της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου υπογράφεται αυτή η συμφωνία. Πόσο πια θα μπορεί να καθυστερήσει κανένας. Αργά με γρήγορα βήματα εναλλάσσονται μεταξύ τους σαν χορό. Ε, αλλά αργό χορό. Ε, η θα γίνει αμοιβή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αλλά αυτό που δεν απαιτεί η συμφωνία είναι η ελευθερία διακίνησης ατόμων, προσώπων. Δηλαδή, το ελεύθερο εμπόριο ε, και η κυκλοφορία, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι πράγματα διαφορετικά. Ορίστε, αυτό λέγαμε κι εμείς ε, ε, για την Βρετανία. Δηλαδή, μπορούμε να καταργήσουμε τους δεδασμούς ε, χωρίς να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Αυτή τη στιγμή επαλευθερώνεται το εμπόριο στις υπηρεσίες. Ε, ταυτόχρονα όμως στη, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να θέσει εμπόδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ε, εξέλθει από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει αυτή την κοινή λογική προ το Ηνωμένο Βασίλειο που δείχνει ήδη στη Σιγκαπούρη. Θα έρθει όμως μια μέρα που ο πρόεδρος του Συμφουλίου, ο κύριο Τάσκ, Τούσκ, θα βρει την θέση που του αξίζει στην κόλαση. Ο κύριο Τούσκ ε, ε, προσπαθεί να δηλητηριάσει την διαδικασία εξώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα το πετύχει. Οπότε συστήνω στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογράψουν μια παρόμοια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αυτή που υπογράφουμε με τη Σιγκαπούρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε μετά ε, ο κύριος, σας ευχαριστούμε για ο κύριος Λαντσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή πόσο αποφελή και ε, θετική μπορεί να είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Σιγκαπούρη. Μου φαίνεται απίστευτο κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μια εμπορική συμφωνία επενδύσεων με κάποιο άλλο μέρο ε, του κόσμου εκτό των σύνορων μα, πάντα είναι υποφελέ αμοιβαίω. Αυτή η συμφωνία ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων σε μια εποχή που έχει ξεπεραστεί από τι εξελίξει τη πραγματικότητα. Η Σιγκαπούρη, όπω φαίνεται από την πρόταση εμπορική συμφωνία, είναι ε, η κοιτίδα τη οικονομία και τη οικονομική ανάπτυξη τη Νοτιοανατολική Ασία. Όμω, συνάδελφοι, την οικονομική ανάπτυξη αυτή θα την ε, καρποθούν άλλοι που δεν είναι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ευνοϊκέ εμπορικέ ρήτρε. Βλέπουμε ότι ε, η Σιγκαπούρη είναι τρίτη χώρα σε προέλευση παραπημένων προϊόντων στον κόσμο βάσει των μελετών καμία καταπολέμηση διαφθορά και η Ιταλική βιομηχανία είναι ένα από τα πρώτα θύματα των παραποιημένων προϊόντων αυτών. Θα ανοίξουμε τι πόρτε σε προϊόντα τα οποία παράγονται με χαμηλό κόστο από τη Μαλαισία, την Κίνα και την ε, Ινδονησία. Και ε, στη Σιγκαπούρη απλώ φτάνουν για το τελευταίο στάδιο επεξεργασία του. Απομένουν πολλέ αμφιβολίε για τι γεωγραφικέ ενδείξει, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Το σύστημα που ισχύει στη Σιγκαπούρη δεν προβλέπει καν μητρό. Εδώ οι γεωγραφικέ ενδείξει ούτε καν αυτομάτω θα προστατεύουν προστατεύονται οι Ευρωπαίοι ελεγκτέ, θα πρέπει αυτονόμω να κινούν τη σχετική διαδικασία. Η Σιγκαπούρη είναι και κέντρο ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών με την αμοιβαία απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ο βασικό σκοπό τη συμφωνία που θέλει να επιτρέψει να παρακάμπτονται ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα θέματα αυτά. Πολλέ ανεξάρτητε ε, ενώσει και οργανώσει ε, τοποθετούν τη Σιγκαπούρη σε, σε έναν μαύρο κατάλογο φορολογικών παραδείσων παγκοσμίω. Ε, και με φορολογικό αποκλεισμό και με μεταφορά κερδών σε πολυεθνικές που έχουν έδρα στις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Ντέιβιτ Μακάλιστερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες μου και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για την διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, η οποία ήδη αναφέρθηκε ότι έχουμε ένα σύστημα που αναπτύχθηκε εδώ και δεκαετίες, ένα σύστημα πολυμερές παγκοσμίου εμπορίου το οποίο απειλείται και αμφισβητεί τις εταιρικές μας σχέσεις και προσπαθούν κάποιοι με προστατευτισμό να υπαναχωρήσουν από τα συμφωνηθέντα. Γι' αυτό λοιπόν η συμφωνία αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή πηγαίνει πέρα από το καθαρά οικονομικό σκέλος είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς τους εταίρους μας ότι θέλουμε ένα πολυμερές σύστημα με κανόνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Γιώχημ Σούστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε περήφανοι ε, για το ότι δεν θέλουμε απλά ελεύθερο εμπόριο, αλλά με βάση τις αξίες. Και οπωσδήποτε αυτό σημαίνει ότι εμείς ε, και οι εταίροι μας έχουμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην κύρωση των συμβάσεων του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η Σιγκαπούρη αρνείται να το κάνει αυτό ο Υπουργός ε, Εμπορίου από ό,τι φαίνεται έχει μια ιδιαίτερως εχθρική στάση. Αντί για συγκεκριμένα ε, χρονοδιαγράμματα, η επιστολή που μας ε, απέφθηναν ε, περιέχει κάποιες γενικολογίες. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους, όχι μόνο για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει μισθολογικό ντάμπινγκ ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι και ζήτημα αξιοπιστίας. Δηλαδή, αν μιλάμε σοβαρά για εμπόριο που βασίζεται σε αξίες, πρέπει να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μπιλ Έθριτς. Σας ευχαριστώ. Πόσο χαίρομαι που σας συναρπάζει μια εμπορική συμφωνία με μια δυναμική χώρα ε, νησιωτική με χαμηλούς φόρους. Συναρπαστικό και σας έχω νέα Υπάρχει και άλλη μια τέτοια χώρα πολύ πιο κοντά ε, με την οποία μπορεί να κάνετε μια συμφωνία όταν ξυπνήσετε βεβαίως. Βεβαίως όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο η Σιγκαπούρη θα ε, μάλλον έχει ήδη πει ότι θέλει να κάνει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί είμαστε δυναμικές ε, οικονομίες που κινούμαστε γρήγορα δεν καθυστερούμε 10 χρόνια και μέχρι να σκόσουμε το ένα πόδι έχει βρωμίσει άλλο. Λοιπόν, Μιλάμε για το εμπόριο, μιλάμε για το πώς θα γίνουμε πλουσιότεροι και θα εμπορευόμαστε προϊόντα και αγαθά. Δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε κανόνες ο ένας στον άλλον και να περνάει μια δεκαετία. Αναμένω λοιπόν τα ίδια συναρπαστικά να ζήσουμε και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας αρέσει πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Κολομπιέ. Η σύναψη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη ε, ε, είναι σαν να βοηθάμε την Κίνα. Ε, το 75% των κατοίκων της Σιγκαπούρης είναι Κινέζοι, οπότε είναι η προφυλακή της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαγωγές της Σιγκαπούρης σε μεγάλο βαθμό είναι κινέζικα προϊόντα, τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί από την Κίνα οικονομία της αγοράς δεν είναι κακό ως ε, έννοια, αλλά ε, το σημαντικό είναι να αποφύγουμε θανατηφόρες ανισορροπίες που μπορούν να καταστρέψουν τις οικονομίες μας. Εκεί δεν έχουν τις προδιαγραφές που έχουμε εμείς, ούτε τους κανόνες που έχουμε εμείς. Πολύ δε περισσότερο που το τραπεζικό του σύστημα είναι αδιαφανές. Αυτά μας δημιουργούν ανησυχίες. Οπότε σας καλούμε να απορρίψετε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να προστατεύσουμε οικονομικά την Ευρώπη και ιδιαίτερως τη Γαλλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος... ναι, ο λόγος του κύριο Σαλαφράνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τους συγητές. Ήδη υπογραμμίστηκε η στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής με τη Σιγκαπούρη είναι ο πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Νοτιοανατολική Ασία και τρίτο εξαγωγέα μετά την Κίνα και την Ιαπωνία από αυτή την περιοχή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα περισσότερο την προσέγγιση ε, ενός ε, ελεύθερου εμπορίου δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες. Οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να είχαν υπογραφεί πιο νωρί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όπως είπε η κυρία Μάλστρομ, πολύ συχνά στον καιρό τη παγκοσμιοποίηση δεν γίνεται λόγος μόνο για εισαγωγέ και εξαγωγές, αλλά για πολύ περίπλοκες αλυσίδες παραγωγής με εισαγωγέ από διάφορα σημεία ε, τα οποία, ε, προϊόντα τα οποία συναρμολογούνται κάπου αλλού κλπ. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. Następnym mówcą jest pani Κέρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Σιγκαπούρη και πολύ σωστά προσπαθούμε να βαθύνουμε τη σχέση μα μαζί τη. Η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει, οι συμφωνίε αυτέ θα αποτελέσουν μοντέλο για άλλε χώρε τη περιοχή. Οι εμπορικέ συμφωνίε όμω από μόνε του δεν χρησιμεύουν αν οι κανόνε οι οποίε διέπουν ωφελούν του λίγου και όχι του πολλού. Θα, ε, η συμφωνία αυτή όμως έχει ένα πλαίσιο κανόνων ε, που όμως βασίστηκαν σε πολιτικές υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής που μπορεί να μην υλοποιηθούν. Δεν θέλω να δοθούν περισσότερα προνόμια σε επιχειρήσεις, σε ανθρώπους όπως ο κύριος Γκουάμ, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιν της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτέλους τελειώνει αυτή η διαδικασία και αύριο θα ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι εδώ και χρόνια έτοιμη η συμφωνία. Ε, αποφασίσαμε όμως να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με βάση αυτή τη συμφωνία ενώπιον του δικαστηρίου. Καμία άλλη συμφωνία δεν έχει εξεταστεί τόσο πολύ από το δικαστήριο όσο αυτή. Και επιτέλου κάναμε με τη Σιγκαπούρη αυτό με το οποίο κάναμε με Καναδά και Ιαπωνία και θέλουμε να κάνουμε και με άλλε χώρε, δηλαδή κανόνε για το παγκόσμιο εμπόριο, έτσι ώστε να μην επικρατεί ο μεγαλύτερο και ισχυρότερο, όπω λένε κάποιοι συνάδελφοι, αλλά να υπάρχουν κανόνε και ένα σαφέ πλαίσιο. Γι' αυτό το ερώτημά μου προ του συναδέλφου που απορρίπτουν αυτή τη συμφωνία είναι τι θα προκύψει καλύτερο αν απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία. Χάνουμε πολλές ευκαιρίες, αφήνουμε σε άλλους την αγορά, χάνουν τζίρο οι εργαζόμενοι μα. Ε, δεν βελτιώνουμε τίποτα εάν καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους να ξανασκεφτούν μέχρι αύριο τις τάσεις τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Σίλβα Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το κοινοβούλιο μας πρέπει να εγκρίνει αμελητή τις τρεις σημαντικές αυτές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη που είναι ε, στο επιτάπητος για την οικονομία μας και για να δικαιωθεί η στατική σημασία της σχέσης με την Σιγκαπούρη. Ε, είναι σημαντικό για την πρόθεση των επενδύσεών μας, διότι είναι ακόμη ένα βήμα για την εκρίζωση των συστημάτων ιδιωτικού δικαίου και έτσι θα, περάσουν θα καταργηθούν τρει ε, διμερεί συμφωνίε που είναι απερχαιωμένε. Επίση, η συμφωνία για τα εμπορικά θέμα γιατί διευκολύνει την εμπορική σχέση μα με ένα σημαντικό εταίρο στην Ανατολική Ασία, προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη και περιέχει συμβαστικέ μάλλον παραχωρήσει τη Σιγκαπούρη, πολύ σημαντικέ, για την κύρωση των ε, συμβάσεων του Διεθνού Οργανισμού Εργασία, του ILO. Επίση, ε, θα εγκρίνουμε ένα προοδευτικό ψήφισμα, όπω αυτό που έχει προτείνει ο συνάδελφό μα Δάβιδ Μάρτιν. Και επίση, χωρί να καθυστερήσουμε, θα πρέπει να εγκρίνουμε και τι τρει αυτέ συμφωνίε. Ευχαριστούμε και τώρα από το ΕΛΚ e ο κύριο Φιέλνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, επιτέλους, έχουμε αυτή τη συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Ε, θα πρέπει να ήταν απλά τα πράγματα, όμως χρειάστηκε μια δεκαετία και δεν έχετε οι Σιγκαπουριανοί. Εμεί στέγαμε. Ε, πολλοί ήταν οι συνάδελφοι εδώ στο σώμα που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την ε, παρακολύσουν, ιδίω ό,τι αφορά τι επενδύσει, τη Συμφωνία για τι Επενδύσει και συνεχίζουν να παρακολύουν. Αυτό έχει βλάψει, έχει θίξει την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Και η Σιγκαπούρη ε, δεν ε, έτυχε δίκαιε μεταχείριση. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι τη συμφωνία αυτή τη θεωρώ καλή. Τη θεωρώ μια πολύ δυναμική οικονομία τη Ανατολική Ασία στη Σιγκαπούρη. Και νομίζω ότι αύριο θα πρέπει να τη δικαιώσουμε. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έγκριση των συμφωνιών αυτών. Ε, υπάρχουν πολλοί εδώ που είναι κατά ε, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Προσπαθούν να παρακολύσουν την πρόοδο της εμπορικής μας πολιτικής ε, με πρόσχημα την Κίνα. Είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ευρεία στήριξη και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στην όλη διαδικασία. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Είμαι Μέλο τη αντιπροσωπεία με ε, των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών ΑΖΕΑΝ. Και θεωρώ ότι οι χώρε αυτέ μπορούν να προσφέρουν πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα την ευκαιρία να, συνετήσω, να συζητήσω τη συμφωνία αυτή με μια σειρά από ε, συνομιλητές της Σιγκαπούρη, με κυβερνητικέ οργανώσεις, εκπροσώπους ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όλοι θέλουν μια ισχυρότερη σχέση συνεργασία, εταιρική σχέση μεταξύ ε, ημών και ημών. Θεωρούμε ότι το Διεθνέ εμπόριο βρίσκεται σε κατάσταση μεταβαλλόμενη οι Ηνωμένε Πολιτείε ξαναγράφουν ε, παλιού κανόνε που ήταν παγιωμένοι. Δεν είναι αξιόπιστο εμπορικό εταίρο. Γνωρίζω πλήρω, ε, έχω πλήρη επενδυνόση μάλλον το γεγονότο ότι κάποιοι συνάδελφοι διστάζουν, ιδίω ε, για το αν θα κυρώσει η Σιγκαπούρη τι συμβάσει του ΑΕΛΟ και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ έχω λάβει εγγυήσει από τον συγγητή David Martin, που έχει κάνει φανταστική δουλειά ω συγγητή και ο οποίο έχει πιέσει του Σιγκαπουριανού να αναγνωρίσουν πολλέ από τι προτεραιότητε μα, με επιστολή εκ μέρου του Πρωθυπουργού να εκφράζει τι δεσμεύσει και τι υποσχέσει του για τι συμβάσει ΑΕΛΟ και με συμπερίληψη δικτών ε, συγκριτική ε, ε, αξιολόγηση για την περιβαλλοντικά Έχω λάβει όλα αυτά και αυτό δεν είναι μόνο για να σας επενέσω, δεν είναι μόνο για σας κέρδο και ένα ένας παραπάνω πόντος Ντέιβιντ, αλλά για ολόκληρη την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κυρία Γκίλ, ο χρόνος σας τελείωσε. Κύριος Βαλέντσα. Βαλένσα. Αύριο θα ψηφίσουμε προκειμένου να διατηρήσουμε το διεθνή, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών και να βελτιώσουμε το, το, την ελευθερία του εμπορίου. Με βάση όμως ε, αρχές, τις συγκεκριμένες αρχές που έχουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ίσους κανόνες, ίσους όρους και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά με περηφάνεια θέτουμε διαγραφές προδιαγραφές και πρότυπα στο, στην παγκόσμια σκηνή. Και οι επιχειρήσεις μας μεγαλώνουν. Οι εμπορικές ε, συμφωνίες ε, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ε, έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο προτιμησιακών συμφωνιών, πάνω από 70 στον κόσμο. Και δημιουργούμε θέσεις εργασία στην Ευρώπη. Και μια ακόμα φορά, οι εμπορικέ συμφωνίε με χώρε όπω η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ εφαρμόζονται μία-μία και μα ωφελούν. Θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτέ τι ευκαιρίες και στο μέλλον. Αύριο ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. pan pan wiceprzewodniczący telika eh, Οι συμφωνίε αυτές είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πρέπει να κλειστεί στα σύνορά τη. Αντιθέτω, θα πρέπει να ανοιχτεί στον κόσμο δυναμικά και δραστήρια προκειμένου να ρυθμίσουμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Αυτή, αυτές οι συμφωνίες ε, συνεργασίας είναι ένα σημαντικό σημείο φετηρίας για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή τόσο σημαντική στον κόσμο όπως είναι η Νοτιοτεολική Ασία. Θα αποτελέσει τη βάση για την βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης, θα ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και θα επιτρέψει την καλύτερη συνεργασία σε μια ευρεία σειρά τομέων. Η... Θα αποτελέσει μοντέλο ε, τέτοιων συμφωνιών, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τα όπλα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, την προστασία του περιβάλλοντος, η διεθνή συμφωνία κλπ. Την ενέργεια, τις μεταφορές, όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, μα ενημέρωσαν ότι έχουμε μείνει 25 λεπτά πίσω από το διαγράμμα μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο καθένα να σέβεται ακριβώ και να τηρεί το χρόνο το οποίο του απονέμεται. Δεν θα επιτρέψω μπλε κάρτε. Οπότε μία ακόμα φορά, καλησπέρα σας, ο κ. Πέτρελ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον David Μάρτιν για την εξαιρετική του έκθεση. Η συνεργασία και η εταιρική σχέση με τη Σιγκαπούρη περιλαμβάνει όχι μόνο την προστασία των επενδύσεων, αλλά μια γενικότερη πολιτική σχέση που θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε πιο εντατικά, πιο στενά και για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ασφάλεια, για την ανάπτυξη κλπ. Οι συμφωνίες αυτές ανοίγουν καινούριε ευκαιρίες συνεργασία και στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και άλλους τύπους συνεργασία μεταξύ αυτών και της υγείας. Η συμφωνία αυτή θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε μαζί τον καρκίνο και μας ανοίγει τα σύνορα όλης της περιοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Η συμφωνία είναι αρκετά ισορροπημένη και εξ όσων γνωρίζω η Σιγκαπούρη έχει δεσμευτεί ότι θα κυρώσει τη συμβάση του αελαιού του δυνατόν. Αλλά αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό είναι η παρακολούθηση των συνεπειών από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονό είναι ότι η Σιγκαπούρη είναι πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά την ε, διαφθορά, δηλαδή θεωρείται μη διαφθαρμένη χώρα, αλλά περιέργως ε, έχει και πολύ ισχυρό τραπεζικό απόρριτο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποια μέτρα για να ισχύουν αυτά για τα κράτη-μέλη. Προσφάτως είχαμε ένα πρωτόκολλο αποφυγής διπλής φορολογίας με την ε, Λετωνία για να ενισχυθούν οι αμοιβέ επενδύσεις. Και βεβαίως δεν ξέρουμε εάν τα ιδιαίτερα δικαιώματα των επενδυτών είναι συμβατά με τα ανθρώπινα και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Βεβαίως πολλά εξαρτώνται εδώ πέρα από την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαιτήσει την εφαρμογή των συμφωνηθένων. Σας ευχαριστώ κύριε Μάμικινς Σδρογεύσκη λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όλη αυτή η υπόθεση ξεκίνησε το 2014 με ένα ερώτημα προς το ΔΕΚ λάβαμε τις απαντήσεις το 2017, τώρα έχουμε 2019 και ε, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ ε, και αυτές ε, περιμένουν την σύναψη νέας συμφωνίας μετά την συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Θα ήθελα να πω πως είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένος για την συμφωνία με τον Καναδά. Κατά την άποψή μου η προστασία των επενδύσεων, η αποφυγή διπλής φορολογίας και η έλλειψη δασμών είναι υποφελής για τους εταίρους μας και για εμάς. Πρέπει να μας χαροποιεί να προσθέσω πως οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε είναι πολύ δυσκίνητες και θέτουν σε κίνδυνο τις δεσμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν να γίνουν ε, πιο γρήγοροι. Σας ευχαριστώ Μπουσό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την Συμφωνία Εταιρικής ε, Σχέσης και συγχαίρω τις διαπραγματευτικές ομάδες. Η Σιγκαπούρη είναι εδώ και καιρό ένας αξιόπιστος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενείται και χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες και βεβαίως ε, έχει τις ίδιες αξίες με εμά για μια ελεύθερη και ανταγωνιστική οικονομία και κράτος δικαίου. Ιδρυτικό μέλος του ΑΖΙΑΝ, μεγάλος κόμβος της ε, περιοχής και εγώ θεωρώ ότι ε, η σχέση αυτή έχει στη βαρύ γεωστρατηγική βάση για την ε, μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αζίαν. Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εξαγωγής ε, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και έτσι θα δώσει μια όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία 550 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Λοιπόν, ε, κλείνει εδώ ο κατάλογος. Ε, πρώτος στον λόγο έχει ο κύριος Πόσπισιλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για εσάς ε, κυρία Επίτροπε επειδή οριστικοποιήσατε αυτήν την συμφωνία. Θα πρέπει να προωθούμε τις αρχές του ελευθερίου εμπορίου ε, σε αντίθεση με την τωρινή Αμερικανική κυβέρνηση. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε τέτοιες ε, συμφωνίες ε, και να μειωθεί ο χρόνος της διαπραγμάτευσης. Έχουν πέρασει σχεδόν 10 χρόνια βεβαίως. Είχε εμπλακεί και το δικαστήριο, αλλά ας σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να υπογράφουμε τέτοιες συμφωνίες πιο γρήγορα. Ελπίζω λοιπόν ε, σιγά σιγά να υπογράψουμε διμερείς συμφωνίες με, τις, με όλες τις χώρες του ΑΖΙΑΝ. Ε, το ελευθερμόριο πρέπει να είναι η ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω πως ε, πιστεύω στο ελεύθερο εμπόριο που θα βασίζεται όμως σε κάποιες κοινέ αξίες και έχουμε κάποιες ε, κοινέ αξίες ε, με την Σιγκαπούρη δηλαδή τις φιλελεύθερες τάσεις, το κράτος δικαίου κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τους ηγητές και τις διαπραγματευτικές ομάδες. Νομίζω ότι βρήκαμε μια ισορροπημένη συμφωνία που αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τις εταιρείε μας, τους πολίτες μας, ε, τα θεσμικά όργανα. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλη συμφωνία θα μπορούσαμε να επιτύχουμε. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη συμφωνία. Απλά θα χάσουμε χρόνο. Οπότε είμαι υπέρ αυτή τη συμφωνία. και σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ενίσχυση των σχέσεων με την ε, Σιγκαπούρη είναι θετική, ανοίγει ένα σημαντικό τομέα εμπορίου και μας δίνει δυνατότητα να με, βελτιώσουμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή. Και βεβαίως ε, υπάρχουν ε, οι κίνδυνοι που είχαμε δει και στην ε, περίπτωση της TTIP, μια μορφή του ISDS, ένα διεθνές ε, δίκαιο το οποίο εγγυάται έναν ιδιαίτερο μηχανισμό επίλυσης διαφορών των επενδυτών με, ξένες, ε, με ξένα κράτη. Θα πρόκειται για ένα μεγάλο λάθος. Ανταυτού θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα υποχρεώνει τις ε, επιχειρήσεις να πληρώνουν για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη και θα αποτελέσει υπόδειγμα για τις συμφωνίες με Κίνα και με άλλες μεγάλες οικονομίες. Σας ευχαριστώ κύριε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγκαμπούρης οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του εμπορίου και αυτό σημαίνει φυσικά αθρώες εισαγωγές φθηνών προϊόντων από την σιγκαπούρη στην ευρωπαϊκή ένωση διότι η σιγκαπούρη στην πράξη είναι το προγεφύρωμα της κίνας. εκεί εισάγονται με τον α ή β τρόπο κινεζικά προϊόντα τα οποία εν συνεχεία θα εισάγονται στην ευρωπαϊκή ένωση. αλλά και όσα κατασκευάζονται στη σιγκαπούρη εκεί ξέρουμε όλοι ότι δεν τηρείται τροπο νομοθεσία. έχουμε ένα κλασικό μισθολογικό ντάμπινγκ. έχουμε επί της ουσίας μια διαδικασία η οποία παραβιάζει οποιαδήποτε έννοια δικαίου εμπορίου είναι μια περιοχή η σιγκαπούρη που αξιοποιείται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της ευρωπαϊκής ένωσης και άλλων χωρών για τη δημιουργία υπερκερδών. είμαι ενάντια φυσικά και στην λογική του isds που υπάρχει που επί του πρακτέου προστατεύει τους επενδυτές εις βάρος των κρατών και τέλος η ευρωπαϊκή ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει ότι στη σιγκαπούρη δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζεται το κράτος δικαίου παραβιάζεται η κάθε δημοκρατική έκφραση και ισχύει ακόμη Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε έτσι με τον ε, κατάλογο. Κυρία Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω μερικές ερωτήσεις. Το ε, κρατικό χρέος εξαιρείται. Ε, είναι σαφές ότι εξαιρείται το κρατικό χρέος από, και η αναδιάρθρωσή του από την προστασία των επενδύσεων. Ε, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών, ο ISDS, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει πλέον. Τον έχουμε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό χάρη στην δική σας παρέμβαση και πιέσεις με ένα, από ναι, ένα νέο, μοντέρνο, σύγχρονο σύστημα το οποίο ο Γενικός Αγγελέας ε, ανέφερε ότι κήρυξε απόλυτα συμμορφούμενο με την ε, ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ε, πλήρης διαφάνεια, διοντολογικός κώδικας, είναι σαφές ποιος μπορεί να προσφέρει και για ποιο λόγο και αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν τις αγορές τους και την οικονομία τους. Ε, δεν, η Σιγκαπούρη δεν αποτελεί φορολογικό παράγοντα, ε, παράδεισο. Ε, είναι προφανές ότι ε, έχουμε δουλειά να κάνουμε για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, η Σιγκαπούρη θα δημιουργήσει ένα μητρό και οι ευρωπαϊκές ε, χώρες θα μπορέσουν να ζητήσουν τη συμπερίληψη των 196 προϊόντων τα οποία είχαμε ήδη απαριθμίσει. Είναι αλήθεια ότι η Σιγκαπούρη θα πρέπει ακόμα να επικυρώσει τρεις συμβάσεις του ILO αλλά γίνεται ήδη πολύ σοβαρή δουλειά στην εσωτερικά στην κυβέρνηση ε, της Σιγκαπούρης σε συνεργασία με τον ILO έτσι ώστε πράγματι να ε, προσαρμοστεί η νομοθεσία της Σιγκαπούρης και να ευθυγραμμιστεί με αυτές τις συμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να επικυρωθούν. Όπως είπατε και εσείς, η κυβέρνηση Σιγκαπούρης έστειλε μια επιστολή για την διαδικασία αυτή. Αν υπερψηφίσετε αύριο με μεγάλη πλειοψηφία, τι συμφωνίε αυτέ, και ελπίζω θα το κάνετε, θα ψηφίσετε υπέρ μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων, ελεύθερων που θα αποτελέσει σημείο αναφορά για πολλέ άλλε μελλοντικέ συμφωνίε με χώρε τη περιοχή αυτή τη Ασία. Είμαστε υπέρ τη Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων, που ακολουθεί την προσέγγιση την οποία εσεί βοηθήσατε να αναπτυχθεί. Θα βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο ε, την τοποθέτηση της ευρύτερης συνεργασίας σε ένα συγκεκριμένο σαφές και σταθερό πλαίσιο σε θέματα όπως ασφάλεια, ε, έρευνα, μέσω της ε, εταιρικής συμφωνίας και θα είναι και η πρώτη συμφωνία την οποία θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την καινούρια σύγχρονη ε, αρχιτεκτονική. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνουμε τον κύκλο των φίλων μας σε χώρες οι οποίες πιστεύουν στην πολυμερή προσέγγιση, που πιστεύουν στους παγκόσμιους κανόνες, χώρες οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα να υπογράφουμε, να συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες που θα είναι ωφέλιμες και προς, για τις δύο πλευρές. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε. Ε... Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να επενέσω το έργο σας και εγώ. Ένας από τους δύο εισηγητές ε, πήρε ε, όλο το χρόνο που χρειαζόταν στην αρχή, που είχε στην αρχή, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτιν. Η κυρία μου απάντησε πολλές από τις ερωτήσεις, αλλά κοιτώ εδώ γύρω και δεν βλέπω κανέναν από αυτούς που επέκριναν τη συμφωνία να είναι εδώ παρόν. Οπότε σε ποιον απαντήσω. Να, να πω όμω, να επαναλάβω ότι σε ό,τι αφορά την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Ανταλλαγών, είναι καλή για την απασχόληση, για τι επενδύσει. Ε, σε ό,τι δεν αφορά τι επενδύσει, είναι η πιο σύγχρονη συμφωνία που έχουμε μέχρι τώρα και θα συμφωνήσω με την Επίτροπο σε αυτό που είπε. Προσπαθούμε να διαβρύνουμε τι σχέσει μα με χώρε οι οποίες σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο που σκεπτόμαστε εμείς. Κάποιες άλλες χώρες προτιμούν τον νόμο της ζούγκλας. Εμείς προτιμούμε κοινού. Πολυμερει κανόνες. Ευχαριστώ. Άρα καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι που δεν είχαν αρκετό χρονομιλίας ε, θα πίστηκαν φαντάζομαι ε, στη διάρκεια των όσων άκουσαν. Ευχαριστώ συνάδελφοι, κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε, η ψηφοφορία είναι αύριο και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποβάθμιση τα δικαιώματα των γυναικών και στη ισότητα των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.